έκθεση της κυρίας Σαχτιέ προχρημεροδότηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων που υποστηρίζονται από την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων. Merci, Monsieur le Président, Madame. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπη. Θα ήθελα να πω καταρχάς ότι είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος για τη δουλειά που κάναμε σε θεσμικό επίπεδο έχει υπάρξει μια πραγματική βούληση και του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Λυπάμαι για την αναχώρηση βέβαια του Συμβουλίου. για να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί και αυτή η πολιτική αποτελεσματικότητα έχει καθορίσει πλέον τη στρατηγική μας. Μπορώ να σας πω λοιπόν Επίτροπε ένα μεγάλο ευχαριστώ Ξεκινήσαμε στις 4 Φεβρουαρίου και αύριο ε, ολοκληρώνουμε τη διαδικασία. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν και πάρα πολλές ε, ευρωπαϊκές αποφάσεις οι οποίες να έχουν προχωρήσει με τέτοια αποτελεσματικότητα. Να ευχαριστήσω επίσης και το σύνολο των σκιωδών. Σιτνένσκα, Λαβάσοβα και Πατρίκ Λοιαρίκ επίσης. Αγαπητοί συνάδελφοι, μπορέσαμε να ξεπεράσουμε τις διαφορές μας, να ενώσουμε τη βούλησή μας γιατί γνωρίζαμε την κατεύθυνση της εργασίας μας. Προσπαθήσαμε να είμαστε αποτελεσματικοί στον τομέα της απασχόλησης των νέων. Η πρωτοβουλία αυτή για την απασχόληση των νέων είναι τελικά το δυσκολότερο, ε, το δυσκολότερο κομμάτι για να βοηθήσουμε τους νέους. Οι περιοχές οι οποίες έχουν τις περισσότερες δυσκολίες, που έχουν τουλάχιστον 25% από 15% σε 25% που είναι σε ανεργία, είναι δύσκολες περιοχές λοιπόν, και το κοινό αυτό των νέων, αυτοί οι νέοι δεν έχουν ε, φυσικά προλάβει να εξειδικευτούν, δεν προλαβαίνουν να μπουν σε θέσεις απασχόλησης, δεν υπάρχει σύμπτωση, δεν υπάρχει αντιστήχηση ανάμεσα στην εκπαίδευσή τους και τις ανάγκες απασχόλησης. Έχουμε δηλαδή να κάνουμε με την πιο σκληρή πλευρά, αν θέλετε, της ε, πορείας αυτής. Ελπίζω να το πετύχουμε. Νομίζω ότι αυτό επικύρωσε εν πολύ στη στρατηγική μας. Σαν εισηγήτρια για τη συγκεκριμένη έκθεση εξέφρασα την επιθυμία ανάμεσα σε όλες τις πολιτικές ομάδες να συμμεριστούμε τον μέγιστο δυνατό αριθμό θεμάτων και θέσεων. Συναντηθήκαμε όσο χρειαζόταν για να ευθυγραμμίσουμε τις πολιτικές μας βουλήσεις με έναν στόχο την επιτυχία των νέων. Λοιπόν, είμαι περήφανη για την Ευρώπη σήμερα. Όχι μόνο πετυχαίνουμε ε, ομόφωνα σχεδόν σε επίπεδο επιτροπής να ανταποκριθούμε σε μια πραγματική εκ των κάτω ανάγκη. Αυτή είναι η Ευρώπη δείχνει η Ευρώπη ότι γνωρίζει τις ανάγκες των νέων. Τα λειτουργικά προγράμματα καθυστέρησαν είναι αλήθεια. Και τι χρειάζονται αυτοί οι νέοι. Αυτό το οποίο χρειάζονται είναι να έχουν στη διάθεσή τους μια σημαντική προχρηματοδότηση. Όταν είπατε ότι αυτό θα περάσει από το 1% στο 30% αυτό σημαίνει ότι η Ευρώπη αναγνωρίζει τις τοπικές ανάγκες. Αυτοί που προωθούν προγράμματα, ιδιαίτερα στις δύσκολες περιοχές, δεν μπορούν να έχουν τις προκαταβολές αυτές στη διάθεσή τους. Οπότε η βοήθεια που δίδουμε είναι ιδιαίτερα καθοριστική. Είναι ένας αγώνας ενάντια στον χρόνο αυτό στον οποίο κάνουμε και ελπίζω να πετύχουμε από κοινού. Θα πρέπει λοιπόν σήμερα για μια ακόμη φορά λέγω να είμαι θα υπερήφανη για την προσπάθεια και αύριο η ψηφοφορία έχει πολύ μεγάλη σημασία. Είναι μια ψηφοφορία μήνυμα έτσι ώστε σε όλα τα κράτη-μέλη να μπορέσουμε να ανασκουμποθούμε και να βοηθήσουμε το πρόγραμμα αυτό για τους νέους. Αυτό χρειαζόμαστε. Το Συμβούλιο τώρα είναι αυτό που θα πρέπει να δώσει τα κίνητρα που απαιτούνται έτσι ώστε οι νέοι να βοηθούν να προχρηματοδότηση την οποία παρέχει η Ένωση πλέον. Ευχαριστούμε πολύ κυρία εισηγήτριά μου Μαρέν Σαρτιέ. Τώρα η Επίτροπος Τίσεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, θέλω να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα την κυρία Μωρέν Σαρτιέ γιατί δίνεται προτεραιότητα στο θέμα αυτό για, καθώς και την ευχαριστώ για τον επικοδομητικό τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε το θέμα. Συγχαίρω το Κοινοβούλιο για την ταχύτατη αυτή συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ μας και με το Συμβούλιο και αυτό το βασικό θέμα υποβοήθησης της απασχόλησης των νέων στην Ένωση. Επίσης παράλληλα θα ήθελα να συγχαρώ τη Λετωνική Προεδρία για την δέσμευσή της και την αφοσίωσή της σε αυτό το θέμα. Πράγμα που δείχνει ότι η προτεραιότητα να αντιμετωπιστεί η ανεργία των νέων στην Ευρώπη είναι προτεραιότητα για, όλους, για όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Δεν πρέπει να χαθεί άλλος χρόνος όσον αφορά την γρήγορη εφαρμογή της πρωτοβουλίας για τους νέους. Ο χρόνος είναι σημαντικό στοιχείο για να λυθεί αυτό το πρόβλημα της ανεργίας τους και πρέπει όλοι να αντιμετωπίσουμε τις ευθύνες και τις δεσμεύσεις μας. Όλοι συλλογικά αυτό κάνουμε προτείνοντας διαπραγματευόμενοι και εγκρίνοντας αυτό το νομοθέτημα τόσο γρήγορα. Η σημερινή πρόταση αφορά την επίλυση ενός προβλήματος που είχαμε ταυτίσει από τα κράτη-μέλη, δηλαδή την παρεμπόδιση της γρήγορης εφαρμογής της πρωτοβουλίας για την ανεργία των νέων και η οποία παρεμποδίζεται από την έλλειψη χρημάτων προτείνουμε το 2015 να αρχίσει προχρηματοδότηση κατά περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό θα βοηθήσει στην επιτάχυνση της εφαρμογής της πρωτοβουλίας και θα έχει επίπτωση στη ζωή περίπου 50.000 νέων ήδη. Είμαστε πεπισμένοι ότι η πρόταση αυτή που είμαι σίγουροι ότι θα εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία αποτελεί ένα σημαντικό κίνητρο για τα κράτη-μέλη για να επιταχύνουν και τα δικά τους προγράμματα και να υποστηρίξουν μαθητείες και θέσεις απασχόλησης για τη συνέχιση της εκπαίδευσης. Κύριοι κυρίες βουλευτέ, σε όλα τα κράτη-μέλη πλέον έχει αρχίσει η εφαρμογή με απτά αποτελέσματα, όπως φαίνεται και από τα παραδείγματα στην ε, έκθεση για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο η εγγύηση αυτή έχει δώσει την όθηση για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και επίσης υπήρξε καταλήτης για τη στήριξη των νέων που μόλις βγαίνουν από τα σχολεία για να βρουν κάποια δουλειά. Και ελπίζουμε ότι έτσι θα επιταχυνθεί περαιτέρω η εφαρμογή λόγω του επίγοντα χαρακτήρα του θέματος. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι η Κομισιόν θέλει να αρχίσει προχρηματοδότηση αμέσως μόλις τεθεί ενισχύει ο τροποποιημένος κανονισμός. Το βασικό θέμα βέβαια είναι η ποιότητα των στηρικτικών μέτρων, των μέτρων στήριξης και επ' αυτού η Κομισιόν θα συνεχίσει να υποπτεύει στενά την εφαρμογή και φυσικά θα σας αναφέρει όπως χρειάζεται, όπως πρέπει. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Εξονόματος της Επιτροπής Πολιτισμού η κυρία Σιλβή Γκυγιόμ έχει το λόγο. Παρακαλώ. Ε, chers collègues, cette proposition vient répondre à une situation que nous avons eue euh, maintes fois. Πολλές φορές ε, κράσαμε τη λύπη μας για την κατάσταση που επικρατεί ως προς την ανεργία των νέων γιατί ακούστηκαν πολλά μέτρα λήψη αλλά δεν απέφεραν αποτελέσματα. Ένας νέος στους πέντε βρίσκεται σε ανανεργία στην Ευρώπη. Είναι δύσκολη λοιπόν η εφαρμογή, ανεπαρκής οι επενδύσεις. Όλα αυτά ε, είναι αρνητικά σημάδια για την εφαρμογή της πρωτοβουλίας των νέων. Εμείς αρνούμαστε να θυσιάσουμε ολόκληρη γενιά. Επομένως το, η πρόταση που έχουμε μπροστά μας είναι απαραίτητη ώστε να υποφεληθούν οι νέοι που έχουν διπλώματα εκείνοι που δεν έχουν και να μπορέσουν να παραμείνουν σε επαφή με τον κόσμο της εργασίας και κυρίως είναι απαραίτητη για να αποφευχθεί η μακροχρόνια ανεργία και οι αρνητικές της συνέπειες. Οι νέοι είναι τα κύρια θύματα της κρίσης που ξέσπασε από το 8 και μετά και κυρίως εκείνοι που δεν έχουν επαρκή διπλώματα ή εκπαίδευση. Οι νέοι με που προέρχονται από τη μετανάστευση αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα μεγάλο πρόβλημα και δεν πρέπει να το παραγνωρίσουμε. Έπρεπε λοιπόν να αντιδράσουμε σύντομα, γρήγορα και αυτό πραγματικά έκανε το Κοινοβούλιο και σα ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ. Τώρα θα ακούσουμε τις πολιτικές ομάδες. Πρώτα απ' όλα η κυρία Λαρακόμη από το ΕΛΚ για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για μια εξαιρετική δουλειά. Η πρόταση αυτή είναι μια εξαιρετική πρόταση και προβλέπει την αύξηση της προχρηματοδότησης των λειτουργικών προγραμμάτων για την πρωτοβουλία για τους νέους η προκαταβολή ενός δις από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το πέρασμα από την προχρηματοδότηση του 1% στο 30% είναι μια ουσιαστική βοήθεια που θα καταστήσει το μέσο αυτό λειτουργικό. Γιατί δυστυχώς τα κράτη-μέλη δεν έχουν προβλέψει ε, εθνικούς πόρους. Η Ευρώπη πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί για να μειώσει την ανεργία και στους νέους. Απευθύνω έκκληση στα κράτη-μέλη και στις περιφέρειες έτσι ώστε να λάβουν υπόψη τους σοβαρά την προτεραιότητα της βοήθειας προς την απασχόληση των νέων. Από τις εμπειρίες τις οποίες ε, είχαμε μέχρι σήμερα βλέπουμε ότι η Ευρώπη είναι ταχύτατη μερικές φορές αντίθετα από ό,τι πιστεύουν ορισμένοι. Το θέμα είναι ότι η εφαρμογή καθυστερεί στα κράτη-μέλη. Σε ορισμένες χώρες το πρόγραμμα αυτό πήγε καλά, σε άλλες χώρες δεν έχει πάει καθόλου καλά. Κλείνω λοιπόν λέγοντας ότι απαιτείται μεγαλύτερη επικοινωνία ανάμεσα στην Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους πολίτες, γιατί πολλές φορές δεν γνωρίζουν τι ευκαιρίες έχουν και τις χάνουν τις ευκαιρίες αυτές. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Κόμη, δέχεστε μία μπλε κάρτα. Κυρία Φρόντε, αν ακούσαμε καλά. Θα ήθελα να ζητήσω από την κυρία Κόμη, μιας και αναφέρθηκε, αναφέρθηκε στο πρόγραμμα εγγύησεων για τους νέους, αν γνωρίζει ότι το ελεγκτικό συνέδριο παρουσίασε μια έκθεση επ' αυτού και να εμείνω σε αυτά τα οποία είπε για την Ιταλία, ότι το πρόγραμμα αυτό δεν απέδωσε τίποτα στη χώρα μου. Πιστεύετε ότι στο μέλλον θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις έτσι ώστε το πρόγραμμα αυτό να καταστεί αποτελεσματικό. Ευχαριστώ τον κύριο Αφρόντε. Ως Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος υπεύθυνη για τα θέματα της νεότητας έχουμε προχωρήσει μαζί με άλλους συναδέλφους σε μια ανάλυση της υπόθεσης αυτή σε επίπεδο ευρωπαϊκό και κυρίως ιταλικό. Στη Λομβαρδία, στην περιοχή μου, το πρόγραμμα της ε, των εγγύσεων για τους νέους είναι το καλύτερο από όλοι στην Ιταλία. Στην Ιταλία γενικά όμως μένουν πολλά να γίνουν. Ο άνεργος μπορεί να είναι κομμουνιστής, φασίστας, σοσιαλιστής, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ο άνθρωπος να βρει δουλειά. Η κυρία Κόμη μπορεί να απαντήσει. Όχι. Ε, ο κύριος Μπενιφέη για τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ πρόεδρε. Είναι εξαιρετική η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το Κοινοβουλίο έχει επιδείξει την απαιτούμενη ευθύνη. Και ήδη αύριο θα ψηφίσουμε. 5 δις προχρηματοδότησης θα τεθούν στη διάθεση των ανέργων νέων. Στη χώρα μου από 5 εκατομμύρια ευρώ θα περάσουμε σε 75 εκατομμύρια διαθεσίμων για τα προγράμματα τα λειτουργικά. Ευχαριστώ την Επίτροπο Τάισεν γιατί μπόρεσε να κατανοήσει το αίτημα και της δικής μας πολιτικής ομάδας που ζητά την αύξηση του ποσοστού προχρηματοδότησης των λειτουργικών προγραμμάτων για να αποφύγουμε τα προβλήματα ρευστότητας των κρατών μελών και των περιφερειών. Η Ευρώπη έκανε αυτό που έπρεπε. Τα κράτη-μέλη τώρα είναι αυτά τα οποία θα πρέπει να αποδείξουν ότι είναι σε θέση να ξεπεράσουν τα γραφειοκρατικά προβλήματα, να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις, και θα πρέπει η προσφορά να είναι ποιοτική και να βοηθήσει την εξέλιξη των νέων με ποιοτικά χαρακτηριστικά. Απαιτείται διαφάνεια, σωστή διαχείριση και εκεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο θα είναι πολύ προσεκτικά. Με τους συναδέλφους της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων προετοιμάζουμε και μια προφορική ερώτηση προς τα κράτη-μέλη για να προκαλέσουμε τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια από πλευράς τους. Πρέπει λοιπόν το συμπληρωματικό αυτό ποσό να μεταφερθεί στα κράτη-μέλη χωρίς καθυστέρηση. Κάθε κυβέρνηση πρέπει να επιδείξει την απαιτούμενη σοβαρότητα. Δεν θα πρέπει να χάσουμε αυτή τη γενιά. Είναι η γενιά μου και πρέπει να βοηθηθεί να βρει το μέλλον της. Έτσι θα ξεπεράσουμε την κρίση και εμείς σαν βουλευτές είναι καθήκον μας να βοηθούμε. Ευχαριστώ πολύ για την ομάδα των συντηρητικών. Η κυρία Γιάννα Ζιτνάνσκα. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλοι γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι να αρχίσουν οι νέοι να δουλεύουν, να μπορούν να είναι ενεργά μέλη της ε, κοινωνίας. Ιδεοδός θα έπρεπε η αγορά εργασίας να μπορεί να τα προσφέρει αυτά χωρίς παρέμβαση, αλλά δεν ζούμε σε ιδεώδη κόσμο, αλλά σε ένα κόσμο εκατοντάδες χιλιάδες άνεργους νέους. Γι' αυτό συμφωνούμε με τους ε, εισηγητές ε, για το ότι πρέπει να βοηθήσουμε τους νέους. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Αλλά αυτό δεν φτάνει. Τώρα πρέπει τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν ε, σωστά τα κονδύλια αυτά. Αλλιώς θα συνεισφέρουν στην περαιτέρω απογοήτευση των νέων. Σας ευχαριστώ για τους φιλελεύθερους η κυρία Ντλαμπάγιοβα. Για δύο λεπτά σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Ευχαριστώ την κυρία Σιγήτρη για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε που απέδειξε πως μπορούμε να αντιδράσουμε ως Ευρώπη. Τώρα ε, πρέπει να αντιδράσουν τα κράτη-μέλη. Σύμφωνα με μια τσεχική εφημερίδα, η Πράγα έχει τη χαμηλότερη ενεργεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση 2,5%. Θαυμάσια νέα, αλλά πρέπει να το δούμε αυτό στο γενικότερο πλαίσιο. Γιατί αν δούμε την ανεργία των νέων, είναι 10%. Βεβαίω ε, είναι πάρα πολύ καλό ποσοστό σε σχέση με την Ήπειρο, όπου έχουν 70% ανεργία των νέων. Γι' αυτό όμως πρέπει ακριβώς να εστιάσουμε στις ε, περιφέρειες που χρειάζονται τη βοήθειά μας. Η πρωτοβουλία αυτή έχει έναν προϋπολογισμό 3,2 δις, ε, εκ των οποίων 1 δισεκατομμύριο θα εκταμιευθεί αμέσως 4 εκατομμύρια για την Τσεχία. Αλλά βεβαίως δουλειές για την νεολαία πρέπει να δημιουργηθούν σύμφωνα με τις ανάγκες της οικονομίας. Γι' αυτό ακριβώς πρέπει να συμπληρωθούν και από εθνικά μέτρα αυτές τις πρωτοβουλίες. Ειδικά η μετάβαση από το σχολείο στην εργασία πρέπει να είναι φυσική και ομαλή. Πρέπει λοιπόν να ευθυγραμμίσουμε τις ανάγκες και τις δεξιότητες με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Πρέπει να στηρίξουμε τις νέες εταιρείες, την μαθητεία, την πρακτική και να κάνουμε περισσότερα για να βοηθήσουμε να αντιμετωπιστούν οι πραγματικές αιτίες της ανεργίας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Για την ε, Γκουε, ο κύριος Λέιερικ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύρια Επίτροπε, κύριε και κύριοι. Είναι επίγον να δοθεί κάποια απάντηση στο δράμα της ανεργίας των νέων και γι' αυτό χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία της προχρηματοδότησης και του άμεσου ξεπλοκαρίσματος ενός δισεκατομμυρίου για την ε, απασχόληση των νέων. Τώρα πρέπει τα κράτη-μέλη να δεσμευτούν και τα χρήματα αυτά να φτάσουν πράγματι στα χέρια των δικαιούχων. Από την άλλη μεριά πρέπει να προσέξουμε το πρόγραμμα αυτό να διαιωνιστεί, να σταθεροποιηθεί ώστε να αυξηθεί όντω η απασχολησιμότητα των νέων. Εγκρίνουμε λοιπόν την έκθεση της κυρίας Μωρέν Σαρτιέ, αλλά γνωρίζουμε ότι είναι πολύ περιορισμένη αυτή η πρόοδος που αντιπροσωπεύει για να αντιμετωπιστούν τα εκατομμύρια των νέων που αυτή τη στιγμή δεν έχουν επαγγελματική εκπαίδευση και δουλειά. Εδώ πρόκειται για για πραγματικό δικαίωμα, δικαίωμα στην εργασία μια Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιμόρφωσης και Ασφάλειας της Απασχόλησης νομίζω ότι θα ήταν επίγον να δημιουργηθεί για να υπάρξει μέλλον για κάθε νέο Ευρωπαίο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Βουλευτά. Εξ ονόματος των Πρασίνων, Ράιντκε. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι και κράτη-μέλη μόνο για δέκα μήνες είμαι βουλευτής και ήδη έχω βαρεθεί με τις ομιλίες για την ανεργία των νέων χωρίς καμία δράση καθώς και γιατί τα κράτη-μέλη δεν παίρνουν σοβαρά τις ευθύνες τους. Όλο τα ίδια λέγουμε. Ίσως να φταίω εγώ, ίσως να είμαι πολύ ανυπόμονη, αλλά έχω ακούσει πάρα πολλές ιστορίες ε, με ανεργία των νέων. Μα για όνομα του Θεού είμαστε στα μέσα του 15. Ξυπνήστε επιτέλους κράτη-μέλη. Κοιμηθήκατε πολύ χρόνο. Το 30% προχρηματοδότησης προτείνει τώρα η Κομισιόν για την Πρωτοβουλία των Νέων είναι ίσως η τελευταία φορά που θα σας ζητήσουμε να ξυπνήσετε. Μετά πρέπει να εφαρμοστεί μια γρήγορη διαδικασία γιατί όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να αντιδράσουμε τώρα Τώρα πρέπει και τα κράτη-μέλη να κάνουν το ίδιο, να χρησιμοποιήσουν τα χρήματα και να φτάσουν αυτά στους νέους. Διότι η δική τους πολιτική ευθύνη είναι. Ευχαριστούμε. Δέχεστε γαλάζια κάρτα από τον κύριο Γιάκοφτσιτς. Ναι. Ορίστε κύριε Γιάκοφτσιτς. Ευχαριστώ που δεχτήκατε τη γαλάζια κάρτα. Θέλω να σας ρωτήσω αν και καταλαβαίνω το θυμό σας, δεν θα συμφωνούσατε ότι η απόφαση αυτή να αυξηθεί προχρηματοδότηση κατά 33% δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αξιόπιστη και ότι η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο έχουν ως προτεραιότητα την προστασία των δικαιωμάτων των ανέργων νέων. Δεν νομίζετε ότι τελικά έχουμε αξιοπιστία. Ορίστε. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Συμφωνώ ότι δεχόμαστε και εμείς αυτή την πρόταση και ότι στο Κοινοβούλιο κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να προωθηθούν τα πράγματα γρήγορα. Τώρα όμως είναι ευθύνη των χωρών μελών να δράσουν γιατί εκείνες έχουν την ευθύνη να χρησιμοποιήσουν τα χρήματα αυτά, να φτάσουν αυτά στους νέους και να μεταφραστούν σε προγράμματα που να είναι χρήσιμα για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων. Ευχαριστώ. Κυρία Ράιντκε, τώρα για την Ευρώπη της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας, η κυρία Λαουρα Αγκαία για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, ευχαριστώ την εισηγήτρια. Συμφωνούμε εδώ πέρα σε αυτή την κατεπίγουσα διαδικασία, αλλά Εμένα μου έρχεται να πω πως η εγχείρηση επέτυχε και ο ασθενής απέθανε. Εγώ είμαι μαθημένη στην ε, αυτοκριτική. Θα μιλήσω για τη χώρα μου λοιπόν, την Ιταλία. Μιλάνε για το να ε, για το πώς θα βρουν τις απαραίτητες πόρους με τρόπο ο οποίος πραγματικά με ντροπιάζει και με ντροπιάζει επίσης το πώς διαχειρίζονται την λεγόμενη εγγύηση της νεολαίας. Μιλάμε για ένα κουτί άδειο το οποίο δεν εκμεταλλεύονται, δεν το έχουν διαφημίσει, δεν το ξέρει ο κόσμος ποιο είναι ε, τα δικαιώματά του και ποιες ευκαιρίες έχουν. Δεν υπήρξε καμία παρακολούθηση, δεν υπήρξε καμία ενημέρωση. Αυτή είναι η αξιολόγηση την οποία πρέπει να κάνω σήμερα. Ντρέπομαι για την ε, χώρα μου η οποία περιγράφηκε από το ελεγκτικό συνέδριο ως μία από τις πέντε χώρες η οποία δεν είχε κανένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα για τους νέους τους. Η Ευρώπη και η χώρα μου πραγματικά αποτυγχάνουν εδώ πέρα και χρεοκοπούν. Σας ευχαριστώ. Δέχεστε μία μπλε κάρτα από τον κύριο Μπονιφέη. Ναι, ωραία. Κύριε Βουλευτά, ευχαριστώ Δεδομένου του ενδιαφέροντος που υπάρχει για αυτήν την συζήτηση υπήρξαν διάφορα σχόλια. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω κυρία Αγκαία γιατί ο σκιώδης εισηγητής για το EFD ε, δεν ήρθε σε κάποιες ε, συναντήσεις και έστελνε τους ε, βοηθούς της. Ε, θα μας βοηθούσε πάρα πολύ στην ε, υιοθέτηση του κειμένου και της επιστολής που αποστήλαμε προς Συμβούλιο και Κομισιόν. Δεν νομίζετε πως ε, αν μια επιτροπή παλεύει μήνες για να βελτιώσει ένα κείμενο αξίζει να αφιερώσετε λίγο χρόνο από το να έρχεστε τώρα μόλις στην Ολομέλεια. Ευχαριστώ τον συνάδελφο, τον Μπραντο Μπενιφέη αλλά ανήκοντας σε μία από τις ε, μικρότερες ομάδες αυτού του Κοινοβουλίου είμαι εισηγήτρια σε δύο άλλες εκθέσεις. Αν ο κύριος Μπενιφέη εργαζόταν με τον ίδιο ζήλο που εργάζομαι εγώ, τότε θα μπορούσε να ασκήσει όση κριτική θέλει. Η κυβέρνηση όμως εδώ πέρα κατασπατάλησε το πρόγραμμα αυτό της εγγύησης για τους νέους και κατασπατάλησε εκατομμύρια ε, ευρώ και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να πούμε. Μάλιστα, έχουμε έναν ενδοϊταλικό ε, διάλογο. Λοιπόν, Μαρούσικ ε, τώρα έχει τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι, πρέπει να καταλάβουμε ότι η ανεργία μια κατηγορία πληθυσμού, στην περίπτωσή μα των νέων, είναι ένα από τα στοιχεία της γενικότερης ανεργίας. Γι' αυτό δεν θα έπρεπε να μαζεύουμε τα σκουπίδια κάτω από το χαλί απλώς για ένα μερικό τμήμα του προβλήματος. Αν χρησιμοποιήσουμε τεχνητό τρόπο για να φέρουμε τους νέους αυτούς στην αγορά εργασίας, αυτό θα μεταφραστεί απλώς σε ακόμα μεγαλύτερη ανεργία μεταξύ άλλων ομάδων του πληθυσμού. Τους ψηλούς, τους κοντούς, τους αριστερόχειρες κτλ. Η ανεργία είναι αποτέλεσμα λανθασμένων θεσμών και δομών πρέπει να μιλήσουμε για τους λόγους, για τη ρίζα του κακού, η οποία είναι αναποτελεσματικό οικονομικό σύστημα. Δεν απασχολούνται από εταιρείε οι άνθρωποι, αλλά από καταναλωτές. Όταν οι καταναλωτές έχουν χρήματα, τα δαπανούν και προσλαμβάνουν ανθρώπους. Ο κύριος Βαντεν Κέντελαρ από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, 7 εκατομμύρια άνεργοι νέοι. Δηλαδή μιλάμε για φοβερά νούμερα και απαράδεκτη κατάσταση. Πλέον έχουμε υποθηκεύσει όχι μόνο το μέλλον τους, αλλά το μέλλον ολόκληρης της Ένωσης. Πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα και να αλλάξουν γρήγορα. Η συμφωνία αυτή είναι μια σημαντική αρχή για να δοθεί μια όθηση και θα πρέπει να δοθεί βάρος ειδικά στις ε, περιοχές οι οποίες πλήττονται περισσότερο. Η ταχύτητα με την οποία Κοινοβούλιο και Συμβούλιο αντιμετώπισαν το θέμα δείχνει πως η Ευρώπη μπορεί να κινηθεί γρήγορα όταν αυτό απαιτείται και είναι πραγματικά μεγάλη στα μεγάλα και σημαντικά. Θα πρέπει λοιπόν ταυτόχρονα να θέσουμε τους απαραίτητους στόχους και με την ευρωπαϊκή προχρηματοδότηση κατά 30% πλέον δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Αυτή βεβαίως η έξτρα προχρηματοδότηση είναι μόνο ένα βήμα γιατί πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση επιγόντως. Θα πρέπει να έχουμε μια πιο μακροπρόθεσμη στρατηγική με δεξιότητες οι οποίες θα ταιριάζουν καλύτερα σε αυτά τα οποία ζητάει η αγορά, με καλύτερες δυνατότητες μαθητείες και βιώσιμε δουλειέ. Έπρεπε λοιπόν να γίνει αυτή η αρχή. Τώρα το μπαλάκι είναι στα κράτη-μέλη. Το σημαντικότερο ερώτημα λοιπόν που πρέπει να θέσουμε σήμερα δεν είναι το τι θα κάνουν τα κράτη-μέλη. Το ερώτημα που πρέπει να απαντήσουμε είναι τι κάνουμε στη συνέχεια. Ο κάθε ε, παίκτη του σκακιού σκέφτεται πολλά θέματα μπροστά. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε και εμεί για να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα. Σα ευχαριστώ η κυρία Στάινρουκ για 1,5 λεπτό. Δυστυχώς σήμερα δεν εορτάζουμε κάποια μεγάλη επιτυχία στην καταπολέμηση της ανεργίας των ε, νέων. Απέχουμε ακόμα έτη φωτός από αυτό. Επιτέλους έχουμε μια πρωτοβουλία σε αυτό το θέμα και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ε, συμμετέχοντες γιατί υπήρξε μια κινητοποίηση γιατί τα τελευταία χρόνια μόνο λόγια είχαμε ο ένας περνούσε τον παπά στον άλλον αλλά δεν κάναμε τίποτα. Οι σοσιαλδημοκράτες είχαν πει πως η καταπολέμηση ανεργίας ε, των νέων δεν αντιμετωπίζεται μέσω της ε, αυστηρής λιτότητας αλλά μέσω μιας ε, κοινής ευρωπαϊκής ανάληψης ευθύνης και δεν χρειάζεται να είναι κανείς μάντης για να καταλάβει πως πρέπει να βοηθήσουμε ακριβώς τα κράτη-μέλη εκείνα τα οποία πλήττονται από την λιτότητα. Χρειάζονται λοιπόν στήριξη και στις σωστές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Η καταπολέμηση της ανεργίας των νέων πρέπει να παραμείνει απόλυτη προτεραιότητα. Το είπατε κυρία Επίτροπο, όχι μόνο στα κράτη-μέλη αλλά και στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και παντού. Και τώρα οι κυβερνήσεις και οι επιχειρήσεις της χώρας θα πρέπει να κάνουν κάτι για τις νέες γενιές που χρειάζονται μια προοπτική και πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια γι' αυτό. Σας ευχαριστώ. Κυρία Στάινρουκ. Τώρα κυρία Μακίντάιρ. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όλοι αναγνωρίζουμε ότι η ανεργία των νέων είναι σοβαρότατο θέμα και υπάρχει τεράστια ανάγκη για δράση. Υποστηρίζω λοιπόν την πρόταση που θέτει στη διάθεση των προγραμμάτων αυτών πιστώσεις για την επιτάχυνση της εφαρμογής τους. Έχω όμως και κάποιες ανησυχίες γιατί η προχρηματοδότηση θα πιέσει οικονομικά το ταμείο αυτό και θα χρειαστούν ε, σε λίγα χρόνια επιπλέον χρήματα για την πρωτοβουλία για τους νέους. Εμείς έχουμε ζητήσει σαν πολιτική ομάδα για δημοσιονομική πειθαρχία και αξιολόγηση εκ των αποτελεσμάτων. Ως εκ τούτου θα πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί σε σχέση με τα αποτελέσματα. Θα πρέπει να συνεργαστούμε με τα κράτη-μέλη για να βρεθούν λύσεις οι οποίες θα ελαφρύνουν τα προβλήματά τους. Συμπληρώνει εθνικά προγράμματα η κυβέρνηση, η δική μου, και στα Ανατολικά Μίλαντς έχουν συγκεκριμένες εταιρικέ μορφές συνεργασίας για έβρεση θέσεων απασχόλησης. Ε, και στα Δυτικά Midlands έχουν ξεκινήσει τα τελευταία πέντε χρόνια 2,5 εκατομμύρια νέες θέσεις μαθητείας για νέους. Η κυρία Ζούμπερ έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η πρωτοβουλία αυτή για την προχρηματοδότηση των προγραμμάτων των νέων είναι κάτι το απαραίτητο. Βέβαια στην αρχή το ποσό αυτό ήταν τόσο χαμηλό που η συγχρηματοδότηση από πλευρά των κρατών μελών δεν ήταν εφικτή. Γιατί οι χώρες αυτές ε, ξέρετε ότι έχουν τεράστια ποσοστά ανεργίας και δεν μπορούσαν να βοηθήσουν. Η πρωτοβουλία αυτή λοιπόν δυστυχώς συνοδεύεται από ένα πολύ χαμηλό προϋπολογισμό και δεν μπορεί να επηρεάσει ιδιαίτερα τα πράγματα και να λύσει τα προβλήματα της ανεργίας των νέων. Γνωρίζουμε ότι στα πλαίσια της εφαρμογής του προγράμματος οι θέσεις απασχόλησης οι οποίες έχουν δημιουργηθεί είναι λιγότερες από τις θέσεις εργασίας τις οποίες καταργούμε μέσω της πολιτικής που ακολουθούμε. Και πολλές φορές τα στάζ και οι προσωρινές θέσεις απασχόλησης αντικαθιστούν τη μόνιμη απασχόληση. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Φουντούλης έχει το λόγο. Ένα λεπτό παρακαλώ λέει ελληνικά ο πρόεδρος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων προσπαθεί να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα που είναι υπαρκτό και ιδιαίτερα έντονο ειδικά σε χώρες όπως η δική μου. για να γίνω πιο συγκεκριμένος στην ελλάδα το ποσοστό ανεργίας των νέων επίσημα προσεγγίζει το 60% ενώ στην πραγματικότητα ίσως να είναι ακόμα μεγαλύτερο. ακόμα χειρότερα δεν προβλέπεται αυτή η κατάσταση να αλλάξει σύντομα παρά τις προσπάθειες που γίνονται τόσο σε εθνικό όσο και σε επίπεδο ένωσης ο λόγος που δεν πιστεύω πως θα αλλάξουν τα πράγματα είναι η λάθος προσέγγιση που έχουμε απέναντι στο πρόβλημα. αντί να επιδιώξουμε τη δημιουργία μόνιμων και αξιοπρεπώς αμοιβόμενων θέσεων εργασίας επικεντρωνόμαστε σε μια αμφιβόλου αξίας επανεκπαίδευση καθώς επίσης και στη δημιουργία προσωρινών και χαμηλά αμοιβόμενων προγραμμάτων απασχόλησης με αυτόν τον τρόπο τα πραγματικά σημαντικά ποσά που δαπανούνται δεν θα έχουν στο τέλος κανένα αποτέλεσμα πέρα από το οικονομικό όφελος ορισμένων που παριστάνουν πως ενδιαφέρονται για τη λύση του προβλήματος της ανεργίας ενώ απλά έχουν βρει ένα ακόμα τρόπο για να απομυζούν χρήματα από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. σας ευχαριστώ. ευχαριστώ. Ε, σας ευχαριστώ. κυρία το σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι θετική η απόφαση της εισηγήτριας, η πρόταση της εισηγήτριας και πρέπει να στηρίξουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αύξηση των προκαταβολών στα προγράμματα που αφορούν τους νέους. Το ένα δις το 2015 αποδεικνύει παρά τους περιορισμούς ότι ο αγώνας κατά της ανεργίας γίνεται με σοβαρό τρόπο. Ε, θα πρέπει τα χρήματα αυτά να χρησιμοποιηθούν με αποτελεσματικό βέβαια τρόπο και γι' αυτό θα παρακολουθήσουμε από πολύ κοντά τον τρόπο που θα δράσουν οι κυβερνήσεις. Εγώ είμαι σε στενή επαφή με τους υπευθύνους στο Υπουργείο Εργασίας και εξετάζουμε τον τρόπο με τον οποίο προετοιμάζονται τα προγράμματα αυτά. Νομίζω ότι η τσεχική δημοκρατία είναι σε θέση να τα εκμεταλλευτεί σωστά, ιδιαίτερα σε περιοχές με υψηλή ανεργία. Πέρα από την Πράγα που έχει χαμηλή ανεργία, έχουμε άλλες περιοχές με ανεργία άνω του 25% στους νέους. Στους νέους μέχρι τα 25%. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να υπάρξει η περισσότερη στήριξη ε, στην επαγγελματική κατάρτιση κυρίως. Πρόκειται για μια επένδυση στο μέλλον των παιδιών μας. Πρόκειται για μια επένδυση η οποία θα δημιουργήσει κίνητρα και θάρρος στους νέους. Η κυρία Ουλφσκοκ έχει το λόγο. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ακούσαμε με πολύ ενδιαφέρον το τι συνέβη στην Ιταλία και σε άλλες χώρες. Να σας πω τι γίνεται στη Σουηδία, όπου υποτίθεται ότι η κατάσταση δεν είναι πάρα πολύ δύσκολη. Παρ' όλα αυτά η ανεργία των νέων είναι αρκετά υψηλή, είναι πολύ υψηλή θα έλεγα και γι' αυτό δόθηκε μεγάλη σημασία στην πρωτοβουλία αυτή για τους νέους. Οι σουηδικές κυβερνήσεις, η προηγούμενη μάλλον σουηδική κυβέρνηση, μείωσε το εύρος των προγραμμάτων αυτών γιατί δεν ήθελε ε, να χρησιμοποιήσει τον εθνικό προϋπολογισμό και προτιμούσε την αναμονή μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Αυτή η στάση, αυτή η νοοτροπία πρέπει να αλλάξει πλέον Υπάρχουν πολλές χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου οι οικονομικές συνθήκες ε, ήταν πραγματικά καταστροφικές και δεν υπήρχε δυνατότητα στήριξης αυτής της πρωτοβουλίας λόγω έλλειψης πιστώσεων. Οι επιπλέον πόροι λοιπόν τώρα μπορούν να λειτουργήσουν θετικά και να κυνηγήσουμε την ανεργία αυτή που χτυπά τους νέους αλλά όταν οι χώρες είναι πολύ φτωχές θα χρησιμοποιήσουν ακόμα καλύτερα αυτή την πρωτοβουλία. Ευχαριστώ πολύ. Ιάν Σάντερ έχει το λόγο. Ενάμιση λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να χαιρετήσω την προσπάθεια την οποία έκανε ο εισηγητής και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι προκαταβολές αυτές, οι προχρηματοδοτήσεις αυτές για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων δεν είναι παρά ένα καλό νέο. Αποδεικνύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν θέλει μπορεί να δράσει γρήγορα και αποτελεσματικά. Τώρα πια ε, το παιχνίδι θα πρέπει να το παίξουν τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα, να ενθαρρύνουν τις διαδικασίες κατάρτισης και μαθητείας να δώσουν, να εμφυσίσουν στους νέους το πνεύμα της επιχειρηματικότητας και να προσαρμόσουν τη διδασκαλία και την παιδαγωγική τους στον νέο ψηφιακό κόσμο. Να επιμείνω τώρα σε ένα επιμέρους θέμα, την κινητικότητα τη διασυνοριακή. Θα επιτρέψει στους νέους να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες τις επαγγελματικές και πέρα από τα κοντινά του σύνορα αυτό περνά και μέσω από την διδασκαλία των ξένων γλωσσών. Δυστυχώς όμως η γαλλική κυβέρνηση θέλει να καταργήσει ε, τα δίγλωσσα σχολεία, κάτι το οποίο είναι κατά της προσπάθειας την οποία κάνουμε εμείς εδώ σήμερα. Η κινητικότητα των νέων περνά και από μια καλύτερη ενημέρωση για την ύπαρξη θέσεων εργασίας στο εξωτερικό και ε, για την αμοιβαία αναγνώριση των διπλωμάτων. Είναι μέτρα μεταξύ τους διαφορετικά αλλά συμπληρωματικά και από κοινού θα καταπολεμήσουμε την ανεργία των νέων. Ευχαριστώ πολύ κυρία Σαντέρ. Η κυρία Μπλινκεβιτσίουτε έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συγχαίρω για την έκθεση και την Κομισιόν που αποφάσισε την αρχή της προχρηματοδότησης γιατί έτσι θα βοηθηθούν τα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της ανεργίας των νέων όσο δυνατόν αποτελεσματικότερα. Οι νέοι χρειάζονται κάποια βοήθεια για να βρουν μια δουλειά, να συνεχίσουν την επιμόρφωσή τους ή τη μαθητεία τους. Σύμφωνα με τις τελευταίες εκθέσεις, λόγω της κρίσης, δεν μπορούν όλα τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν την πρωτοβουλία για την νεολαία και γι' αυτό η πρόταση αυτή είναι σημαντικό θετικό βήμα και επένδυση προς τους νέους, για τους νέους. Κατά την εφαρμογή των μέτρων της πρωτοβουλίας για την νεολαία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία σε εκείνους που έχουν χαμηλότερη επιμόρφωση ή στους ασθενέστερους που έχουν κάποια ασθένεια. Δηλαδή. Θα ήθελα να τονίσω ότι η μακροχρόνια ανεργία των νέων έχει πολύ αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία και μπορεί να έχει αρνητική επίπτωση και πάνω στους ίδιους τους νέους ας πούμε μπορεί να αναπτύξουν υγειονομικά προβλήματα ή διανοητικά προβλήματα ή να καταλήξουν εγκληματίες. Ευχαριστούμε. Ε, ο κύριος Λόπες, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς θα ήθελα να καλωσορίσω την Επίτροπο έτσι ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες ε, ε, προχρηματοδότησης στις χώρες που έχουν ανάγκη ε, από την προώθηση των προγραμμάτων αυτών. Θα ήθελα να θυμίσω ότι τα κράτη-μέλη, αυτά τα οποία έχουν τα πιο σοβαρά προβλήματα με την ανεργία των νέων, έχουν και τα πιο σοβαρά προβλήματα με το θέμα του ελλείμματος. Ε, το θέμα, η προσπάθεια την οποία κάνουμε είναι μια μικρή προσπάθεια χωρίς αποτελέσματα που θα γλυκάνει λίγο την κατάσταση προσωρινά. Το θέμα είναι να αλλάξουμε τις πολιτικές μας στο Καδίς, στο νότο της Ευρώπης, είναι υπόδειγμα του τι συμβαίνει στο νότο της Ευρώπης. Πραγματικά υπάρχει μια τεράστια, ένα τεράστιο ποσοστό ανεργίας. Έχουν δημιουργηθεί κατεπίγουσες καταστάσεις τις οποίες καλούμεθα και σαν Ευρωπαϊκή Ένωση και σαν κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Λόπες. Φτάσαμε τώρα στη διαδικασία Catch από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια, του και τις εισηγητές και την Επίτροπο για την έκθεση αυτή. Γιατί είναι κάτι το ιδιαίτερα σημαντικό για τους νέους της Ευρώπης να στηριχθούν δηλαδή και να έχουν την απαραίτητη κατάρτιση για να μπορέσουν να απασχοληθούν το γεγονός ότι λέτε πως θα πρέπει να υπάρξει αυτή η προχρηματοδότηση ε, και να δημιουργηθούν οι απαραίτητε δομέ είναι κάτι το ιδιαίτερα ενθαρρυντικό όπως και το ότι λέτε ότι θα παρακολουθείτε την πρόοδο και θα ενημερώνετε τακτικά το Κοινοβούλιο. Γιατί νομίζω πως είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξοδευτούν σωστά αυτά τα λεφτά δηλαδή να υπάρξει η σωστή η κατάρτιση στο χώρο εργασίας γιατί συχνά ε, εκπαιδεύαμε τους νέους και όχι τόσο νέους σε καριέρες ε, και δεξιότητες που δεν χρειάζονται. Πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό το θέμα. Thank you. Σας ευχαριστώ. κύριος Νεγκρέσκου έχει τώρα το λόγο. Μικρόφωνο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εφαρμογή αυτού του σχεδίου. Μιλάμε για 7 εκατομμύρια ένεργους νέους, 7 εκατομμύρια μοίρες ανθρώπων. Δεν είναι λίγα πράγματα. Ένα δισεκατομμύριο προχρηματοδότηση για την καταπολέμηση της ανεργίας είναι σημαντικό, αλλά πρέπει να συμπληρωθεί και με άλλα μέτρα. Χαίρομαι που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δείχνει πως μπορεί να κινηθεί γρήγορα για να καταπολεμήσει την ανεργία και πρόκειται για ένα θετικό μήνυμα και θα ήθελα τα κράτη-μέλη να ανταποκριθούν θετικά. και θα ήθελα επίση τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν τα απαραίτητα εφαρμοστικά μέτρα γιατί η Ρουμανία ήταν ένα από τα πρώτα πιλωτικά κράτη. Για να συμβεί όμω αυτό θα πρέπει να δοθούν τα περαιτέρω κονδυλία σε συγκεκριμένα έργα για να βοηθηθούν οι νέοι. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μαριάς έχει το λόγο. Η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων διαθέτει μόνο 6 δισεκατομμύρια ευρώ τη στιγμή που έχουμε πάνω από 5 εκατομμύρια ανέργους νέους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τη στιγμή που ο Ντράγκη διαθέτει 1,13 ευρώ για αγορά κρατικών ομολόγων όλων των κρατών της Ευρωζώνης πλην Ελλάδας και Κύπρου. Επομένως απαιτείται άμεσα μια γενναία αύξηση του ποσού για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων η ανεργία των νέων στην ελλάδα είναι 51,7 σε πολύ υψηλά επίπεδα είναι η ανεργία των νέων και σε ισπανία και πορτογαλία. ταυτόχρονα η μη αποδοτική χρήση της πρωτοβουλίας στις χώρες του ευρωπαϊκού νότου συνίσταται στην έλλειψη των δημοσίων πόρων που χρειάζονται για να δρομολογηθούν έργα που προσφέρουν νέες θέσεις εργασίας πρακτικής άσκησης και κατάρτισης. ταυτόχρονα λόγω των μνημονιακών περικοπών η ελλάδα έχει τις μεγαλύτερες δυσκολίες όσον αφορά την έβρεση συγχρηματοδότησης πολύ περισσότερο τώρα που ο ντράγκη και η παρέα του στην ΕΚΤ έχουν επιβάλει πιστωτική ασφυξία στην ελλάδα. γι' αυτό χρειάζονται ρυθμίσεις που να διευκολύνουν την απορρόφηση των κονδυλίων της πρωτοβουλίας στην ελλάδα και στις χώρες που τέθηκαν σε μνημόνια. ευχαριστώ. ευχαριστώ. Do accept blue card? Δέχεστε μια γαλάζια κάρτα από τον κύριο Νοβακόφ. Ορίστε κύριε Νοβακόφ μου. господин Благодаря и за това, че приехте карта. важно е Κύριε Πρόεδρε, πράγματι είναι πολύ σημαντικό να αυξηθεί η προχρηματοδότηση για τα προγράμματα προώθησης, αντιμετώπισης της ανεργίας των νέων. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε τις μεταρρυθμίσεις και τις επενδύσεις παράλληλα. Δεν μπορούμε μονομερός να πετύχουμε τον στόχο της καταπολέμησης της ανεργίας των νέων. Υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ χωρών μελών προς αυτό και είναι δύσκολο να απορροφηθεί πολλές φορές η, διαθε... η χρηματοδότηση που διαθέτουμε. Γι' αυτό πρέπει και τα κράτη-μέλη να δεσμευθούν ακόμη περισσότερο για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης για τους νέους. Οι προσπάθειες των χωρών μελών πρέπει να έχουν σαν στόχο την εφαρμογή των χρηματοδοτήσεων και μεταρρυθμίσεων. Τι φρονείτε για τις μεταρρυθμίσεις. Ε, Μάριας, παρακαλώ. Να ευχαριστήσω τον κύριο συνάδελφο και να πω το εξής. Αυτή τη στιγμή για να υπάρξει η συγχρηματοδότηση από πλευράς Ελλάδος χρειάζονται κεφάλαια. Όταν όμως λόγω του μνημονίου έχουν μειωθεί οι δημόσιες επενδύσεις δεν υπάρχουν τα κεφάλαια αυτά ούτως ώστε από ελληνικής πλευράς να γίνει η συγχρηματοδότηση για να έχουμε τα αποτελεσματικά τα αποτελέσματα που χρειάζονται σε σχέση με την συγκεκριμένη πρωτοβουλία. πολύ περισσότερο όταν υπάρχει πιστωτική ασφυξία στις ελληνικές τράπεζες από την πλευρά της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας που πλέον δεν δίνει ούτε ένα ευρώ στην πράξη στις ελληνικές τράπεζες για να μπορέσουν να κάνουν επενδύσεις. άρα λοιπόν για την ελλάδα τουλάχιστον αυτό είναι το βασικό στοιχείο το οποίο πρέπει να λάβετε υπόψη. Ευχαριστώ. Eh, Τώρα η κυρία Μπιλμπάου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να υποστηρίξω την αλλαγή αυτή του κανονισμού έτσι ώστε να στηριχθεί η ανεργία των νέων είναι μια καθοριστική προτεραιότητα για μας. Θα πρέπει να υπάρξει μια ουσιαστική ανάλυση βέβαια των λόγων για τους οποίους τα κράτη-μέλη δεν μπόρεσαν να παρουσιάσουν τα λειτουργικά προγράμματα. Το πρόβλημα είναι πολλές φορές ότι τα κράτη έχουν την τάση να συγκεντρώνουν τα προγράμματα αυτά και να αφαιρούν τις αρμοδιότητες των περιφερειακών οργάνων που είναι σε θέση να τονώσουν την οικονομία, είναι πολύ κοντά στην σωστή κλίμακα για να πετύχουν τις απαιτούμενες εταιρικές συνεργασίες με τον ιδιωτικό τομέα. Για να αποφύγουμε λοιπόν τέτοιου είδους προβλήματα στο μέλλον θα ήθελα να μας πείτε αν θα κάνετε μια προσεκτική ανάλυση των δράσεων των κυβερνήσεων. Σας ευχαριστώ πολύ. Και η κυρία Λόπες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι δεν είμαστε κατά του προγράμματος των εγγύησεων για τους νέους, αλλά δεν συμμεριζόμεθα τον τρόπο που εφαρμόζεται και ιδιαίτερα στην Ισπανία. Η προχρηματοδότηση είναι κάτι το θετικό, αλλά δεν είναι το κεντρικό πρόβλημα αντίθετα με τις άλλες πολιτικές που επηρεάζουν αρνητικά την απασχόληση των νέων. Τα μέτρα αυτά έχουν δυστυχώς οδηγήσει στην επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας και έχουν απομακρύνει τους νέους από την θέση εργασίας. Με τα μέτρα αυτά δεν διασφαλίζεται η συνέχεια στην θέση εργασίας, η ποιοτική απασχόληση και η σωστή κατάρτιση στο εσωτερικό της απασχόλησης. Αυτά τα προγράμματα θα λειτουργήσουν περιοριστικά θα έλεγα, περιθωριακά και μάλιστα μας προειδοποιεί και το ελεγκτικό συνέδριο για πιθανή στρεβλή χρήση αυτών των προγραμμάτων. Το θέμα είναι να προστατευθούν οι κοινωνικές παροχές και οι μισθοί των εργαζομένων. Ο κύριος Βάλλη έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα εδώ να θέσω ένα θέμα στην Επίτροπο. Θα ήθελα όλα αυτά τα προγράμματα τα οποία αφορούν την απασχόληση των νέων να προσθέτουν, να τα προσφέρουν θέμενη αξία. Δυστυχώς ε, στην δική μου χώρα ο Πρωθυπουργός ότι πετύχαμε τεράστια νίκη ε, με 1,5 δις που οποία πήραμε και τελικά δημιουργήσαμε 12.000 ε, θέσεις ε, απασχόλησης για τους νέους ενώ ήταν 400 τόσοι χιλιάδες οι άνεργοι νέοι. Λοιπόν πρέπει να αλλάξει η στάση αυτή της Ιταλικής κυβέρνησης γιατί αλλιώς η κοινή γνώμη ευρωπαϊκή θα επιδείξει πολύ σκεπτικισμό. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε και κύριοι. Δεδομένη τη κρίσιμη κατάσταση των νέων στην Ευρώπη, η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που στόχο έχει την προχρηματοδότηση τη ε, πρωτοβουλία αυτή μα δίνει δυνατότητα να βελτιώσουμε την κατάσταση. Χαίρομαστε ιδιαίτερα για το ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη αποφάσισαν να εγκρίνουν την πρόταση αυτή χωρί ε, παίρντε τροπολογίε, έτσι ώστε να εκτομιευθούν γρήγορα τα κονδύλια. Η κυρία ε, η δουλειά της κυρίας Μονές Αρτιέ και λοιπόν θα βοηθήσει πάρα πολύ. Όμως δεν αντιμετωπίζουμε τα βασικά προβλήματα των κρατών μελών. Δεν υπάρχει επαρκής εφαρμογή από την αρχή της ε, πρωτοβουλίας αυτής ε, και αντιλαμβανόμαστε πως ε, ο χρόνος εδώ πέρα είναι κρίσιμος παράγοντας ειδικά για όσους είναι ανεργοί εδώ και καιρό και έχουν φοβερές δυσκολίες στο να ξαναμπούν στην αγορά εργασίας και ε, πλησιάζουν πλέον το όριο της ε, φτώχειας και εκεί πέρα πλέον τα πράγματα δυσκολεύουν ε, πάρα πολύ όσον αφορά την επανείσοδο στην αγορά εργασίας. Γι' αυτό ακριβώς η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο πρέπει να ασκήσουν πίεση στα κρατη Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ιβάν Γιάκοβτσιτς. Σας ευχαριστώ. Πρόκειται για μια εξαιρετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θεωρώ πως ε, είναι θετική είδηση για όλους τους νέους ε, στην Ευρώπη γιατί αναγνωρίστηκε αυτό το οποίο ζητούσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το οποίο έχει υποβάλει αυτή την πρόταση για αύξηση της προχρηματοδότησης στο 33% της ε, εγγύησης για την νεολαία. Ήταν κάτι το οποίο περιμέναμε εδώ και καιρό και με τον τρόπο αυτό, κυρία Επίτροπε, θα δείξουμε την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί έτσι ακριβώς μπορούμε να δείξουμε ότι ενδιαφερόμαστε για την επίλυση αυτού του ζητήματος, ειδικά στην ε, Νότια Ευρώπη. Τι ε, πρέπει να γίνει τώρα. Αυτό το οποίο μένει να γίνει είναι ίσως ε, να ενισχυθεί ο αδύναμος κρίκος, δηλαδή τα κράτη-μέλη. Πρέπει λοιπόν να επαγρυπνείτε για να μην υποχωρήσει η αξιοπιστία μας. Σας ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής ο κύριος Αντρέι Νόβακοφ. Благодаря, господин председател. Както казах и преди малко, безспорно 30%... Κύριε Πρόεδρε, είπα και πριν ότι η αύξηση 30% της προχρηματοδότησης των προγραμμάτων για την πρωτοβουλία απασχόλησης των νέων είναι πολύ καλή πρόταση και χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό. Όμως πρέπει να γίνει κάτι παραπάνω και για την επικοινωνία που θα συνοδεύει αυτή την πρωτοβουλία. Πρέπει επίσης να θυμίσουμε το σημαντικό ρόλο που παίζουν οι τοπικές και περιφερειακές αρχές ώστε αυτή η πληροφόρηση και η επικοινωνία να φτάσει μέχρι τους νέους. Γι' αυτό ελπίζω οι χώρες μέλη και οι τοπικές και περιφερειακές αρχές θα κάνουν ό,τι μπορούν για να αυξήσουν τις δυνατότητες τους και να κάνουν παράλληλα τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών απασχόλησης. Έτσι θα μπορούσαμε να διευκολύνουμε την πρόσβαση των νέων στην αγορά εργασίας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Τελείωσε η διαδικασία και της Και δίνω τον λόγο στην Αντιπρόεδρο Τάισεν για την Κομισιόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, σας ευχαριστώ για την στήριξη που επέδειξε ολόκληρο το Κοινοβούλιο στην ε, πρωτοβουλία αυτή και ελπίζω όταν αύριο υπερψηφίσετε αυτή την ε, πρωτοβουλία να ακολουθήσει και το Συμβούλιο και τον Μάιο να περάσουμε σε πληρωμή αυτής ε, της, και εκταμείευση του ποσοστού αυτού της προχρηματοδότησης. Βεβαίως είχαμε και τις διάφορες επιφυλάξεις και φόβους που ακούστηκαν. Γι' αυτό αρχές ε, του 2016 θα γίνει μια συνολική αξιολόγηση για την αποτελεσματικότητα, για τον αντίκτυπο των ε, πραγμάτων ε, αυτών και συγκεκριμένα για την πρωτοβουλία για την απασχόληση της ε, νεολαίας. για την πραγματοποίηση, όπως είπαμε, αυτής της εγγύησης προς τους νέους. Επίσης, θα δώσουμε την βοήθεια στα κράτη-μέλη στις περιφέρειες εκείνες οι οποίες το επιθυμούν. Ένα ερώτημα το οποίο τέθη είναι εάν αρκούν αυτά. Οπωσδήποτε όχι. Αν επαρκεί ο ίδιος ο προϋπολογισμός αυτός για να δημιουργήσουμε όλες τις δουλειές που χρειάζονται, όχι. Προφανώς όχι. Με αυτά τα μέτρα δεν γίνεται. Γι' αυτό ακριβώς έχουμε και άλλα ταμεία ε, που θα χρησιμοποιήσουμε και γνωρίζουμε πως πάρα πολλές χώρες και περιφέρειες πραγματικά είχαν πρόβλημα για να ξεκινήσουν τη χρηματοδότηση κάποιων ε, έργων. Γι' αυτό ακριβώς έφυγε αυτό το εμπόδιο από την ε, μέση. Έχουμε και τα κονδύλια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, του Περιφερειακού Ταμείου, έχουμε το EASY, το πρόγραμμα απασχόλησης και κοινωνικής καινοτομίας και το Erasmus Plus και άλλα προγράμματα. Και όσον αφορά την πολιτική μας βεβαίως δεν αρκούν αυτά. Πρόκειται για ζήτημα προσφοράς και ζήτησης, ε, το ξέρετε αυτό το πράγμα. Γι' αυτό ακριβώς αυτή η Κομισιόν αποδίδει ιδιαίτερο βάρος στην βιώσιμη ανάπτυξη, στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Γι' αυτό ακριβώς μιλάμε για πρωτοβουλίες για να βοηθήσουμε και τους άνεργους για να αυξηθεί και ε, ο σεβασμός των οποίων έχει και απολαμβάνει η επαγγελματική κατάρτιση και άλλα τέτοια πράγματα. Επίσης θα πρέπει να δούμε και το πακέτο επενδύσεων υπ' αυτό το πρίσμα. Γιατί αν ο καθένας αναλάβει τις ευθύνες του τότε μπορούμε να κάνουμε ε, περισσότερα πράγματα και να δώσουμε πρόπτικη στους νέους. Και νομίζω πως έτσι μπορούμε να συνεισφέρουμε και εμείς. Και θα ήθελα και πάλι να σας ευχαριστήσω και να συγχαρώ για την ταχύτητα με την οποία εγκρίθηκε αυτό το Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περνάμε τώρα στην εισηγήτρια, την κυρία Μόνη Σαρτιέ. Euh, Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, θα ήθελα να σας συγχαρώ για τον τρόπο με τον οποίο με τον κανονισμό αυτό συμβάλλεται μαζί με όλους μας τους συναδέλφους στην άρση αυτού του αντιεξόδου που υπήρξε για τη χρηματοδότηση. Το φραγμός αυτός δεν είχε μπορέσει μέχρι τώρα να υπερβληθεί και είναι φανερό ότι η Ευρώπη τουλάχιστον γνωρίζει πια ποιο είναι το πρόβλημα. Κατά την αυριανή ψηφοφορία δεν πρέπει να κάνουμε λάθος συνάδελφοι. Συμφωνούμε επί της ουσίας. Η προχρηματοδότηση αυτή θα συμβάλλει στην επίλυση του προβλήματος της ανεργίας των νέων. Δεν θα τα λύσει όλα βέβαια, το είπε και η κυρία Επίτροπος. Εάν όμως έχουμε μεγάλη πλειοψηφία αύριο τότε θα δείξουμε στο σύνολο των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων ότι έχουμε την απέτηση να αναλάβουν δέσμευση ώστε η πολιτική αυτή να πετύχει. Όχι για να δοξαστούν σε εισαγωγικά αλλά διότι είναι απαραίτητο να αρχίσουν ευρωπαϊκά προγράμματα υπέρ της απασχόλησης των νέων. Αύριο λοιπόν η ψηφοφορία μας και η απέτησή μας αυτή θα φανούν και για τα κράτη-μέλη. Τρίτο θέμα που θέλω να δείξω. Κυρία Επίτροπε, καταλάβατε μάλλον ότι εμείς δεν θα καταλήψουμε τη μάχη. Δηλαδή, η όλη αυτή η εργασία που κάναμε από κοινού για να επιτευχθεί αυτή η προχρηματοδότηση θέλουμε να καταλήξει σε απτά αποτελέσματα τα οποία θα υπάρξουν μόνο αν τα προγράμματα που θα υποπληθούν θα είναι ποιοτικά. Θέλουμε δε και έκθεση αναφορά εποπτεία μαζί με την Επιτροπή, με την και την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων για να γνωρίζουμε ότι υπήρξε αποτέλεσμα των δεσμεύσεών μας κυρία Επίτροπέ μου είμαστε απολύτως δεσμευμένοι επ' αυτού παρακαλώ να καταλήξετε κυρία μου οι μερικοί συνάδελφοι που λένε ότι η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων δεν αρκεί αυτοί θα έπρεπε να ξέρουν ότι έχουμε και άλλα εργαλεία την εγγύηση της νεολαίας και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο που στόχος τους είναι ακριβώς ένας από τους στόχους τους να επανέλθουν οι νέοι στην εργασία, στην απασχόληση. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε κυρία μου. Τελείωσε.